presela. Take your seat. We can start. Καθίστε παρακαλώ στις θέσεις να αρχίσουμε. Βρέθηκε. Όσοι θέλετε να ψηφίσετε, καθίστε. We will start with a small announcement. Θα αρχίσουμε με μία σύντομη ανακοίνωση, γι' αυτό σας παρακαλώ καθίστε. So, Σας παρακαλώ καθίστε. Συνάδελφοι, θα αρχίσουμε με μία ανακοίνωση. Στα τσεχικά, γι' αυτό σας παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Σήμερα διανύουμε την έκτη επέτειο των τρομακρατικών βομβιστικών, της τρομοκρατικής βομβιστικής επίθεσης στο ε, μετρό του Λονδίνου που σκότωσε 52 ανθρώπους και τραυμάτισε 800. Θυμόμαστε πολύ καλά τι συνέβη στις 7 Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο. Πρόκειται για ένα γεγονός που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Σήμερα ιδιαίτερα σκεφτόμαστε τις οικογένειες και φίλους των θυμάτων αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Η βομβιστική επίθεση του Λονδίνου ήταν μία από τις χειρότερες που διεπράχθη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θα ήθελα να υπογραμμίσω προς τους βομβιστές και τους τρομοκράτες ότι ό,τι και να κάνουν δεν θα πετύχουν τους στόχους τους γιατί προσδίδουμε μεγάλη αξία σε κάθε ανθρώπινη ζωή. Žádný terorista či teroristický útok καμία τρομοκρατική δραστηριότητα δεν θα μπορέσει να μειώσει ή να καταστρέψει την πίστη μας σε, στις ανθρώπινες αξίες και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η τρομοκρατία αποτελεί επίθεση προς όλους, μία επίθεση στον ε, δημοκρατικό ιστό της κοινωνίας δεν δικαιολογείται. Η Ευρώπη πάντα θα την καταπολεμήσει. Γι' αυτό θα ήθελα να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή παρακαλώ.